ψυχούν τέτοια ίδια φαινόμενα να μη σε κατανοούν όταν μιλάς τη γλώσσα σου. Αυτά παρακαλώ για τα πρακτικά. Σας ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Λόκεγκαρτ και καταγράφουμε ε, τα λεγόμενά σας. Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα αλλά νομίζω πως εσείς μας διαφωτίσετε για το ποια είναι η θέση σας και θα φαίνεται με σωστό τρόπο στα πρακτικά. Για να ψηφίσουμε λοιπόν την έκθεση Μπαλζάνη Φερνάντες ε, να σας πω πως θα ψηφίσουμε στις 12 και για την έκθεση Μπέγκε η ψηφοφορία θα λάβει χώρα ε, το Νοέμβριο. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε εδώ λοιπόν την έκθεση Γκρέσελ Ριμπελίνη που είναι σχετικά ε, με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης. Η κυρία Γκλέσσερ έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί επέτροποι, η απλούσταυση είναι πολύ δύσκολη σε ορισμένε περιπτώσει. Όσοι εισηγητέ, καταθέσαμε πολλέ ε, τροπολογίε για την ενοποίηση των ε, ε, προβλημάτων και για την επίλυση των προβλημάτων στα ταμεία χωρίς ε, αντίκτυπο στα έξοδα του προσωπικού. Προσπαθήσαμε να μάθουμε από τα λάθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τώρα. Θέλουμε ενιαίους κανόνες προκειμένου να πάρει ένα τέλος αυτή η ποικιλία κανονισμών και θέλουμε πιο πολύ διαφάνεια στον προπολογισμό από ό,τι ως τώρα. Αυτό αποτελεί επίσης ένα μεγάλο βήμα προς την απλούστευση. Να σας ευχαριστήσω όλους όσοι ε, συμβάλλαν τον συνεισηγητή καταρχάς, τα μέλη της ομάδας εργασίας, τους ε, συναδέλφους, τους υπαλλήλους ε, εδώ, αλλά και στην Επιτροπή που μας βοήθησαν. Να βοηθήσω επίσης και τον Κρίστιαν Ζίχελ, ο οποίος ε, είναι ο βοηθός μου και απέκτησε μόλις μωρό. Συγχαρητήρια. Θα ήθελα να πω και να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσει την, ε, τον δρόμο που ξεκίνησε για την απλούστευση. Θα ήταν πραγματικά μεγάλο βήμα αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον οίκο τη, ε, ενιαίου ε, κανόνε. Αυτό θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη συμβολή προ την απλούστευση. Σήμερα ψηφίζουμε το, την έκθεση, τη τροπολογία όχι το ψήφισμα, γιατί ξεκίνησαν συζητήσεις, ε, φιλικές συζητήσεις με το Συμβούλιο και θέλουμε να συνεχιστούν αυτές οι φιλικές συζητήσεις. Σήμερα θα ψηφίσουμε αυτά που δεν πέρασαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να σας πω ότι δεχτήκαμε κάποιες τροπολογίες ως βάση για την, ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας καλέσω για τα χρηματοδοτικά μέσα που για πρώτη φορά γίνεται ορισμός των project bonds να σας καλέσω να περάσουν αυτές οι τροπολογίες γιατί θεωρώ ότι αν υπάρχει μια δέσμευση για την κρίση των χρηματοδοτικών μέσων σε ό,τι αφορά βάση, βάση μάλλον τομέων είναι προς το συμφέρον μας. Θέλουμε οι αρμόδιες, οι επιτροπές ε, να συζητήσουν για την χρήση των χρηματοδοτικών μέσων και να μπορούν να έχουν ε, να ακούσουν τη φωνή τους. και έγινε και προφορική τροπολογία για την ε, τροπολογία 273 όπου τονίζεται ότι θέλουμε να προβλέψουμε μία τομεακή βάση. Να σας ε, προειδοποιήσω σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες 271 278. Ορίζουμε την ανώτατη ευθύνη με τα λεφτά του φορολογούμενου. Θα πρέπει σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο για τα χρήματα του φορολογούμενου, να τον περιορίσουμε κατά το δυνατόν. Αυτό το οφείλουμε στον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Δημιουργούμε λοιπόν μια υποχρέωση αναφοράς από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και θεωρώ ότι αυτά τα οφείλουμε και αυτά στον φορολογούμενο θέλουμε να δούμε πώς θα πάει δύο-τρία χρόνια αυτό το μέσο και να δούμε ποιες λύσεις, ποια συμπεράσματα θα εξαγάγουμε. Θέλουμε δημοσίευση της νομικής μορφής των μέσων ε, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό θα συμβάλλει στην διαφάνεια και θα μπορέσουμε έτσι να ελέγχουμε αυτά που αποφασίσαμε. Καλό θα ήταν αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάνει από μόνη της τις προτάσεις. Επειδή δεν τις έκανε η Επιτροπή πρέπει να τις κάνουμε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ να τις υπερψηφίσει η πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι και πάλι σας ευχαριστώ και χαίρομαι ιδιαίτερα που και στις μελλοντικές συζητήσεις με το Συμβούλιο θεωρώ ότι βρισκόμαστε στον καλό δρόμο, σε καλό δρόμο και σαφώς και θα βρούμε λύσεις σε πολύ σύνθετα νομικά προβλήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκρέσλη. Θα ήθελα να σας πω πως έχουμε κοντά μας σήμερα μία αντιπροσωπεία από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, Ισλανδία, Λιχτεστάν και Νορβηγία.